Λοιπόν, καταληκτικά τέλος της συζήτησης και θα ψηφίσουμε αργότερα σήμερα. Περνάμε στο επόμενο θέμα, κατάσταση στο Τζιμπουτί. Θα δώσω το λόγο για 1,5 λεπτό στην κυρία Ριβαζή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτό το οποίο συμβαίνει στο Τζιμπουτί εδώ και αρκετά χρόνια είναι πολύ ανησυχητικό τα τελευταία γεγονότα μας κάνουν να ανησυχούμε περισσότερο. Αφού άλλαξε το Σύνταγμα για να είναι για τέταρτη φορά υποψήφιος, ο Πρόεδρος επέβαλε μέτρα ελευθεροκτώνα μη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, βία εις βάρος των γυναικών. Το μόνο που μας θυμίζει ότι το Τζιμπουτί είναι δημοκρατία είναι οι τακτικές εκλογές. Οι εκλογές όμως αυτές είναι τέτοιες που ε, τα επίπεδα, τα ψήφου τα οποία παίρνει, τα ποσοστά ο πρόεδρος φτάνει σε δυσθεώρητα ύψη συστηματικά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν συνιστά την δημιουργία μιας ανεξάρτητης εκλογικής επιτροπής. Η γεωγραφία του Τζιμπουτή καθιστά τη χώρα αυτή στρατηγική σημασία και η Γαλλία έχει εγκαταστήσει εκεί την βασική της στρατιωτική βάση στο εξωτερικό. Εν μέρη υπεύθυνη για την κατάσταση είναι η Γαλλία αλλά και άλλες χώρες, η Ιαπωνία, οι Ηνωμένε Πολιτείε και η Κίνα τώρα έχει στρατιωτική βάση στο Τζιμπουτί. Η Ευρώπη πρέπει να δράσει, αλλά και όλες οι χώρες που έχουν εκεί στρατιωτικές βάσεις, έτσι ώστε να μην υπερασπίζονται αυστηρά τα δικαιώματά τους και να σταματήσουν πλέον να είναι υποκριτές. Κοράω ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το Τζιμπούτι είναι το παράδειγμα θα έλεγα της αδυναμίας την οποία έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της εξωτερικής βοήθειας για τη συνεργασία. Το μοναδικό όπλο το οποίο έχουμε για να ζητήσουμε από την ύπατη εκπρόσωπο να κάνει κάτι για το Τζιμπουτί είναι αυτό που κάνουμε σήμερα. Ο χρυσός του Τζιμπουτί είναι η στρατηγική του θέση μετά από τις στρατιωτικές επενδύσεις. Αυτό που μας έλειπε είναι η Κίνα η οποία όμως επένδυσε 80 εκατομμύρια δολάρια και έφτιαξε μια στρατιωτική βάση για 10.000 Κινέζους στρατιώτες. Στο Τζιμπουτί παρά την μεγάλη παρουσία των ξένων στρατιωτών και Ευρωπαίων τα ανθρώπινα δικαιώματα παραβιάζονται συστηματικά εις βάρος των κατοίκων της χώρας. Πρέπει να ζητήσουμε επίσης και από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο να δει τι γίνεται στο Τζιμπουτί για να δούμε αν οι επιθέσεις εις βάρος των τοπικών πληθυσμών μπορεί να θεωρηθούν ως εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Σας ευχαριστώ, μιλήσατε πάρα πολύ καλά αυτή τη φορά. Ο κύριος Τάνοκα ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, ενώ η Σομαλία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τον τζιχαρισμό και την ε, πειρατεία και η Ερυθρέα συνεχίζει τα 30 χρόνια βαρβαρικού καθεστώτος, το Τζιμπούτι δυστυχώ και αυτό είναι ένα κομμάτι αυτής της τριλογίας με τον πρόεδρο Βουέλα, ο οποίος ξεκίνησε την τέταρτη θητεία του μετά από το 87% που πήρε στις εκλογές υποτίθεται, είναι πολύ δύσκολο να περιμένει κανείς μεταρρυθμίσεις και αλλαγή του αυταρχικού του καθεστώτος είδαμε πέρσι να γίνεται μια επίθεση της αστυνομία κατά του ε, γενικού, ε, του ηγέτη του κόμματος της αντιπολίτευσης. Ακολούθησε μια σφαγή όπου σκοτώθηκαν 37 άτομα την ίδια μέρα από τις αρχές. Αυτό είναι ακόμα μια τραγωδία που δείχνει τον βίο και ομό χαρακτήρα της κυβέρνησης του Τσιμπούτη. Υπάρχει μια κουλτούρα καταστολής για τους αγωνιστές των ανθρωπινών δικαιωμάτων και των δημοσιογράφων. Εμεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ασκήσουμε περισσότερη πίεση στην κυβέρνηση του Τζιμπουτή να εφαρμόσει το πλαίσιο πολιτική μεταρρύθμιση που υπεγράφει το 2015 ω σημείο κίνηση για το μέλλον και τη βελτίωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε αυτή τη μικρή αλλά όμορφη χώρα. Παντσέρη. Ευχαριστώ. Στην Αφρική υπάρχουν πολλά πολιτικά καθεστώτα στα οποία η λειτουργία του κράτους γίνεται σε ένα πλαίσιο δυναστικό-οικογενειακό. Στην ουσία την εξουσία έχουν στα πλαίσια της νεποτιστικής αντίληψης του καθεστώτος ε, τα παιδιά και τα ανήψια του Προέδρου. Το μεγαλύτερο τμήμα του πληθυσμού ζει κάτω από συνθήκες φτώχειας ακραίας και υπάρχουν και πάρα πολλοί πρόσφυγες από την Ιεμένη, την Ερυθρέα και τη Σομαλία. Υπάρχουν ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδιαίτερα το νομικά κατώτερο καθεστώς των γυναικών, όπως επίσης και το κρατικό μονοπόλιο στην ενημέρωση. Οι καταγγελίες εις βάρος λοιπόν του Προέδρου Γουέλε, οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να εξετάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να κινηθεί προς την κατεύθυνση αυτή το ταχύτερο δυνατόν. Η κυρία Βευζά ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Επί τη βάση των αναφορών πολλών διπλωματών και ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται εκεί και σε σχέση με τις στρατιωτικές βάσεις που εξαπλώνται στο Τζιμπουτί. Το Τζιμπουτί είναι όαση σταθερότητα. Η πραγματικότητα είναι ακριβώ το αντίθετο. Αυτή τη στιγμή πλήττεται από την οικονομική υπανάπτυξη, από την ένδια η οποία έχει εξαπλωθεί παντού και από την πολιτική καταπίεση. Με το ψήφισμα αυτό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλουμε να βοηθήσουμε και να συγχαρούμε και αυτούς που συνέβαλαν στο ψήφισμα αυτό. Θέλουμε να καταγγείλουμε την κατάστολη που έγινε μετά την ε, ε, σφαγή του World στο το Δεκέμβριο του 2015 και να υποστηρίξουμε αυτούς οι οποίοι έχουν τολμήσει να καταγγείλουν αυτά τα γεγονότα. Πρέπει να σταματήσει και αυτή η φενάκη ε, εκλογικής διαδικασίας που έγινε τον Απρίλιο. Όλοι αυτοί που ξεπερνάνε το 80% σε εκλογική υποστήριξη, αυτά είναι πράγματα μαγειρεμένα. Ακόμα και η Αφρικανική ε, Ένωση θεώρησε ότι υπήρξαν κάποιες ατασταλίες σε αυτές τις εκλογές. Πρέπει να υποστηρίξω και τη φωνή των θαραλέων γυναικών του Τζιμπουτή που έκαναν απεργία πείνα για να καταδείξουν του βιασμού το, του ε, οποίου υπέστησαν από τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων. Χρειάζεται μια διεθνή ανεξάρτητη έρευνα για τα θέματα αυτά και είναι απαραίτητο να μπορέσουμε να δείξουμε όλη την αλήθεια για αυτά που γίνονται στο Τζιμπουτή. Κύριε Γκαμπριέλ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η εταιρική σχέση που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση με το Τζιμπουτί είναι σημαντική ιδίως μέσα στο περιφερειακό πλαίσιο του, κέρα, του κέρατος της Αφρικής σε ό,τι αφορά την ασφάλεια και τον αγώνα κατά της πειρατείας. Γι' αυτό η υποβάθμιση του πολιτικού κλίματος στο Τζιμπουτί, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε αποσταθεροποίηση της χώρας και της περιοχής, μας ανησυχεί τα μάλα σήμερα. Τρία σχόλια. Πρώτα απ' όλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ενθαρρύνει τι αρχέ του Τζιμπουτή να εξασφαλίσουν το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το κράτο δικαίου και τη δημοκρατία. Και επίση να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία στα θέματα αυτά στο εθνικό ενδεικτικό σχέδιο. Δεύτερο, για λόγου αξιοπιστία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι απαραίτητο εμεί να εστιάσουμε στα πιο προβληματικά στοιχεία και να μην χαθούμε σε πολυλογίε για διάφορα θέματα. Το Τζιμπουτί είναι και μια κόλαση για τα ε, είναι μια, ε, ένας χώρος όπου γίνονται, αναγνωρίζονται περισσότερο τα δικαιώματα γυναικών από ότι άλλες περιοχές στην περιοχή. Αυτό δεν είναι το πιο κατεπήγον θέμα. Επίσης θα πρέπει να υπάρξει και μια τακτική διαδικασία για την καταγραφή των παραβιάσεων. Θέλουμε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες και να κάνει το ρόλο της η δικαιοσύνη, αλλά εμείς δεν μπορούμε να καταδικάσουμε από έξω. Ευχαριστώ πάρα πολύ αυτούς που είχαν την επικοδομητική στάση στα ψηφίσματα. Ο κύριος Νάρτ. Δεν τον βλέπω όμως. Προχωρούμε στις ομάδες. Ο κύριος Πόσπιελ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πικροτώ θερμός το ψήφισμα αυτό ως αντίδραση εκλογής του Απριλίου. Για τέταρτη φορά ο πρόεδρος Γκουέλε κέρδισε τις εκλογές και θεωρώ ότι είναι και το πρόσωπο κλειδί αυτός που είναι υπεύθυνο για την τραγωδία ε, σήμερα στο Τζιμπουτί. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό το ψήφισμα στο οποίο ζητούμε ε, να επαληθευθεί, ε, να επαληθευθούν τα αποτελέσματα αυτών των εκλογών που ξέρουμε ότι ακόμα πριν γίνει καταμέτρηση ο πρόεδρος και επίχερε τις της νίκης. Θα πρέπει να παληθευτεί λοιπόν κατά πόσον αυτό το ποσοστό μπορεί να είναι το πραγματικό αποτέλεσμα των εκλογών. Άκρα η φτώχεια, ε, πάρα πολύ κακή κατάσταση των γυναικών, καταστολή ε, της αντιπολίτευσης, ε, δεν υπάρχει δυνατότητα χειραγώγηση των γυναικών. Γι' αυτό και στηρίζω αυτό το ψήφισμα. Πρόεδρος, κύριε Νάρτ, μια και ήρθατε, θέλετε μήπως τώρα να πάρετε το λόγο, να ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε ήθιστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να γίνονται δηλώσεις ε, και καταδίκες που είναι μόνο ρητορικέ για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε πάρα πολλές περιοχές του κόσμου. Το Τζιμπουτί δεν είναι μόνο ένα μέρος που είναι συνήθις η παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά έχει και ευρωπαϊκά στρατεύματα στο έδαφος του. Και από τις βάσεις αυτές ε, λέμε και ε, το κάνουμε, ότι προσπίσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα με την επιχείρηση Αταλάντη ε, συγκεκριμένα. Όμως δεν αρκούν τα ε, λόγια. Πρέπει να πάμε και στα έργα. Θα πρέπει λοιπόν με βάση και το συγκεκριμένο άρθρο της Συμφωνίας του Κοτονού να ζητήσουμε από την κυβέρνηση του Κοτονού να αλλάξει την κατάσταση. Και ευχαριστώ. Η κυρία Ρενά τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα μιλήσω μονάχα για τις γυναίκες του Τζιμπουτί που είχα την ευκαιρία να τις συναντήσω και οι οποίες ήταν θύματα βιασμών. Βιασμών από τους στρατιωτικούς του Τζιμπουτί. Οι γυναίκες αυτές ζητούν απλώς το δικαίωμά τους, το δικαίωμα στη δικαιοσύνη, στην ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Μου μίλησαν πολλοί συνάδελφοι για την κατάσταση για το Τζιμπουτί, παρότι είναι σημαντικό εταίρο στην περιοχή αυτή της Αφρικής, του κέρατος της Αφρικής αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει ατιμορρησία για του δράστε κατά των γυναικών ή οποιοδήποτε άλλο. Θα πρέπει να γίνουν σεβαστά τα πολιτικά δικαιώματα, το δικαίωμα στην ελευθερία έκφραση, το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια, το δικαίωμα στη ζωή απλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Κέλλη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Δυστυχώς έχουμε ξαναδεί το ίδιο έργο και σε πολλά άλλα μέρη. Αυτά που γίνονται στο Τζιμπούτι έχουν γίνει και σε πολλές άλλες περιοχές του κόσμου. Οι ηγέτες θέλουν να παραμείνουν στην εξουσία, χρησιμοποιούν κάθε μέσο, μετέρχονται κάθε τέχνασμα, χρησιμοποιούν το στρατό για να ελέγχει την αντιπολίτευση, δεν επιτρέπουν καμία μορφή ανθρώπινων δικαιωμάτων, καταστέλνουν όλους ιδίως τις γυναίκες, όλα αυτά που γνωρίζουμε και από άλλες περιοχές έχουν γίνει και στο Τζιμπούτι. από το 1999 και την ανάληψη εξουσίας από τον πρόεδρο τον Τωρινό, εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση δίνουμε 105, έχουμε, έχουμε δώσει 105 εκατομμύρια ευρώ στη χώρα αυτή υπό μορφή βοήθειας. Πρέπει να τα επανεξετάσουμε όλα αυτά και θα πρέπει να περιμένουμε, να δούμε τουλάχιστον ότι υπάρχουν, ότι θα λάβουν χώρα ανοιχτές και ελεύθερες εκλογές στη χώρα αυτή. Ο κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η δημοκρατία του Τζιμπουτή βρίσκεται σε μια περιοχή κρίσης. Αυτά τα οποία συμβαίνουν στο κέρας της Αφρικής έχουν άμεσες επιπτώσεις σε όλη την Ευρώπη. Η τρομοκρατία, καταστολή, ε, καταστροφή των κρατικών δομών, όλα αυτά οδηγούν σε κύματα προσφύγων τα οποία έρχονται στην Ευρώπη. Η δημοκρατία του Τζιπλουτή είναι η μικρότερη περιοχή της ε, περιοχής αυτής και θα μπορούσε να είναι μια νησίδα σταθερότητος, ένα υπόδειγμα για όλη αυτή την περιοχή. Η Ευρώπη θεωρεί ότι η χώρα αυτή είναι πολύ σημαντική και την υποστηρίζει αλλά οι εξελίξει οι οποίε ε, αναφέρθηκαν και σήμερα μα οδηγούν σε μεγάλε ανησυχίε. Υπάρχει παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι δεν είναι ανοιχτέ και ελεύθερε οι εκλογέ, όλα αυτά πρέπει να μα οδηγήσουν σε μια κριτική αντιμετώπιση και επομένω δεν πρέπει να μιλάμε μονάχα για τι εξελίξει στην χώρα αυτή, αλλά θα πρέπει να αντλήσουμε και τα απαραίτητα συμπεράσματα σε σχέση με τη δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Περνάω στη διαδικασία Catch the Και δίνω το λόγο στον κύριο Πόλτσακ. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο κυρία Πρόεδρε. Όπως ε, και στην προηγούμενη συζήτηση που είχαμε για την Κάμπη, και στην περίπτωση του Τσιμποτή πρέπει να ε, διαδηλώσουμε την αντίθεσή μας ε, και τον αποτροπιασμό μας για την καταστολή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν ξέρω μήπως είναι πολιτική παράδοση στο Τζιμπουτέ ένας πρόεδρος 20 ε, ετών να δέχεται έναν άλλο, ο οποίος ακολουθεί και την ίδια παράδοση τελικά, αλλά αυτό δεν θα πρέπει εμείς να το υποστηρίξουμε και συμφωνώ με τον κύριο Κέλλη. Όπως και στην περίπτωση της Κάμπια, έτσι και εδώ θα πρέπει να δούμε τι αναπτυξιακή βοήθεια χορηγούμε στη χώρα αυτή γιατί νομίζω ότι αυτά τα 185 ε, εκατομμύρια είναι πάρα πολλά και αν η χώρα δεν μπορεί να πληρεί ούτε τις στοιχειώδεις ε, προϋποθέσεις για την προστασία των δικαιωμάτων ε, θα πρέπει ίσως να επανεξετάσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Μάης. Το Τζιμπουτί παρά το γεγονός ότι κατοικείται από περίπου 864.000 κατοίκους και έχει μικρή έκταση και καθόλου φυσικούς πόρους αποτελεί σημαντική βάση για τις ξένες στρατιωτικές δυνάμεις το τζιμπουτί χαρακτηρίζεται από υψηλή ανεργία και εκτεταμένη φτώχεια ενώ αποτελεί και σημείο διέλευσης για χιλιάδες αφρικανούς μετανάστες. παράλληλα η κυβέρνηση της χώρας ευθύνεται για πολλές περιπτώσεις παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. συγκεκριμένα στις εκλογές του 2013 η κυβέρνηση κατέστηλε βία τις διαδηλώσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης με αποτέλεσμα να υπάρξουν αρκετοί νεκροί. επειδή οι διαδηλωτές αμφισβήτησαν την νομιμότητα των εκλογών για τον λόγο αυτό υπήρξαν μαζικές συλλήψεις και καταγγελίες στη συνέχεια για υπόπτους θανάτους βασανιστήρια και εξαφανίσεις. δεδομένου ότι οι γυναίκες στο τζιμπούτι έρχονται αντιμέτωπες με διάφορες μορφές βίας και οι περιπτώσεις ανελευθερίας του λόγου είναι αρκετές θα πρέπει να υπάρξει πίεση της ευρωπαϊκής ένωσης ώστε να σταματήσει η καταπίεση των δικαιωμάτων στη χώρα. το τζιμπούτι έχει προσυπογράψει τη διεθνή σύμβαση για οικονομικά και πολιτιστικά δικαιώματα του οηε και θα πρέπει να την τηρήσει. ευχαριστώ. Ήταν ο Καστάλντο. Ευχαριστώ. Το Τζιμπουτί είναι μια μικρή χώρα, αλλά ο πρόεδρος Γελέ έχει δημιουργήσει μια ισχυρή δικτατορία με νεποτισμό, διαφθορά. Οι εκλογές είναι ένα ανέκδοτο. Οι αυθαίρετες συλλήψεις, τα βασανιστήρια, η βία είναι καθημερινότητα. Ηνωμένε Πολιτείε, Ιαπωνία, Κίνα κατανοούν τη στρατηγική σημασία και έχουν δημιουργήσει στρατιωτικές βάσεις. Το πλαίσιο είναι ε, θα έλεγα το περιφερειακό εξαιρετικά άσχημο εμείς λοιπόν πρέπει να πούμε όχι, το ψήφισμά μας είναι ένα πρώτο βήμα. Ο εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου πρέπει να προχωρήσει σε έρευνες εις βάρος του Τζιμπουτή και θα πρέπει επίσης να λειτουργήσει και το άρθρο 8 της Συμφωνίας του Κοτονού. Δεν μπορούμε να στηρίζουμε ένα καθιστό το οποίο τραυματίζει με τέτοιο τρόπο τον πληθυσμό του. Η στρατηγική θέση του Τζιμπουτή δεν δικαιολογεί την σιωπή μας. Καλημέρα Πρόεδρε. Νομίζω ότι για μια ακόμη φορά δεν μιλάμε για την ουσία. Υπάρχουν χώρες που έχουν δικτάτορες, απαράδεκτες καταστάσεις, ελλείψεις δημοκρατίας και το θέμα είναι βέβαια τι γινόταν στο παρελθόν, ήταν καλύτερα στο παρελθόν. Βέβαια εδώ εμείς στην Ευρώπη, στην Ιαπωνία, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Κίνα εποφελούμεθα από την κατάσταση. Και τελικά ποιο είναι ο καρπός αυτής της προσπάθειας αυτού του αποτελέσματος είναι ότι ε, δεν έγινε και τίποτα. Θυμάστε την Αραβική Άνοιξη, μας είχαν ζαλίσει τότε και στην ουσία καταλήγουμε στο να λέμε σήμερα ότι οι Αφρικανοί θέλουν τους δικτάτορες διότι η δημοκρατία στην Αφρική δεν πάει καθόλου καλά. Κλείνουμε το Κατστιάι λέει η πρόεδρος. Σας ευχαριστώ. Δίνω το λόγο. Έχετε το λόγο. Κάποιος έχει ζητήσει το λόγο μια στιγμή. Η κυρία Κιέγκε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εμείς ε, θα εκφράσουμε την ανησυχία μας ε, για αυτούς οι οποίοι προσπαθούν μέσα από τον Τζιμπουτί να ξεφύγουν από τους πολέμους και από την πείνα και να προσπαθήσουν να φτάσουν είτε στη Βόρεια Αφρική είτε στην Αραβική Χερσόνησο. Θα πρέπει λοιπόν η κυβέρνηση του Τζιμπουτί να διασφαλίσει την ασφάλεια αυτών οι οποίοι προσπαθούν να ξεφύγουν και σε νομικό επίπεδο παίρνοντας μέτρα εις βάρος των εμπόρων ε, της ανθρώπινης αγωνίας. Γίνονται τεράστιες τραγωδίες σαν για αυτές τις οποίες βιώνουμε στη Μεσόγειο και για τις οποίες αποσιωπούμε θα έλεγα τα πραγματικότητα για το τι πραγματικά συμβαίνει στον κόλπο του Αντένα. Υπάρχουν εγκληματικά δίκτυα λοιπόν, υπάρχει σώματεμπορία, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε ποιοι κερδίζουν από αυτό και σε τοπικό επίπεδο γιατί οι πρόσφυγες είναι τα εύκολα θύματα όπως πάντα. Η Επίτροπος ε, Γιώραβα. Έντιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Τζιμπούτι έχουν μια μακρά σχέση και Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί το Τζιμπούτι ένα σημαντικό εταίρο. Το Τζιμπούτι έχει υποστηρίξει τοπικές και περιφερειακές ε, πρωτοβουλίες και δίδει στα θέματα αποστολέ αποστολές της ε, Αφρικανικής Ένωσης στη Σομαλία που είναι και το κλειδί στον αγώνα κατά της Al-Shabaab και για την εξασφάλιση της πολιτικής διαδικασίας της Σομαλίας. Σε εσωτερικό επίπεδο η ανάπτυξη η εξέλιξη μάλλον των κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Τζιμπουτί είναι κάτι το οποίο μα ανησυχεί. Οι ακτιβιστέ ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοσιογράφοι έχουν υποστεί παρενόχληση και καταστολή και ο πολιτικό χώρο τη αντιπολίτευση έχει συρρυκνωθεί μετά από τι προεδρικέ εκλογέ τη 8η Απριλίου 2016. Σε όλη τη διάρκεια τη προεκλογική περίοδου, μέλη και υποστηριχτέ τη αντιπολίτευση έχουν κρατηθεί, ε, συλληφθεί και κρατηθεί χωρίς κατηγορίες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολούθησε αυτές τις εξελίξεις και έχει εκφράσει την ανησυχία της σε διάφορα επίπεδα. Στις 21 Δεκεμβρίου του 2015 η αστυνομία ε, διέλυσε μια θρησκευτική τελετή κοντά στην πρωτεύουσα του Τζιμπουτή. Η παρέμβαση των αστυνομικών δυνάμεων οδήγησαν σε κάποιους θανάτους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εκδώσει μια δήλωση ζητώντας διευκρίνηση για τα γεγονότα αυτά και για την τιμωρία των δραστών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδικάζει τις βίες αυτές ενέργειες, θεωρεί <clears throat> χρειάζεται μια διεθνής έρευνα για τα θέματα αυτά και είναι υψής της σημασίας. Και επομένως χαίρεται και για την ε, μεσολάβηση του υπάτου του εκπροσώπου για τα ανθρώπινα δικαιώματα του ΟΗΕ που θα είναι στο Τζιμπουτή αυτή τη βδομάδα και που η παρουσία του επιτρέψει τη διευκρίνηση των θεμάτων αυτών σε σχέση με τις πρόσφατες προεδρικέ προεδρικές ε, ε, εκλογές το να υπάρξει ένας κατάλογος <clears throat> αναλυτικός για τα αποτελέσματα σε κάθε εκλογικό τμήμα θα είχε αυξήσει και την εμπιστοσύνη στην ακεραιότητα των αποτελεσμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά να εφαρμοστεί πλήρω η συμφωνία πλαίσιο για τι πολιτικέ και θεσμικέ αλλαγέ που έχει συμφωνηθεί μεταξύ τη κυβέρνηση του Τζιμπουτή και τη αντιπολίτευση στο τέλο του 2014. Αλλά αυτή η διαδικασία έχει τελματώσει από πέρσι. Πρέπει να γίνουν αυτές οι προσπάθειες σε μια διαδικασία δημοκρατικοποίησης στο Τζιμπουτή η δημοκρατικοποίηση και τα θέματα διακυβέρνησης και ο μεγαλύτερος σεβασμός για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί η εσωτερική σταθερότητα του Ζιμπουτή σε μια περιοχή η οποία χαρακτηρίζεται από συγκρούσεις και από ένδια. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να ενθαρρύνει όλες τις πολιτικές δυνάμεις του Τζιμπούτι να ξαναρχίσουν τον πολιτικό διάλογο για να μπορέσουν να προχωρήσουν σε πολιτικές μεταρρυθμίσεις, να βελτιώσουν την διακυβέρνηση και να τεθεί ένα τέρμα στην, ε, στις εντάσεις που έχει γνωρίσει η χώρα τα προηγούμενα χρόνια. Για το θέμα που έθεσε η κυρία Αρένα, ποια είναι η θέση της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τις γυναίκες της, ε, του Τζιμπουτή που έχουν ξεκινήσει απεργία πείνα για να καταγίνουν του διασμού που υπέστησαν από το στρατό της, του Τζιμπουτή. Θέλω να σα διαβεβαιώσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει παρακολουθήσει από πολύ κοντά το θέμα αυτό θεωρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι πρέπει να γίνει μια έρευνα για να διακριβώσει τι έχει γίνει και να έλθουν ενώπιον της δικαιοσύνης οι δράστες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να συνεργαστεί με όλους τους εμπλεκομένους για να βελτιωθεί η κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Έχουμε έξι ψηφίσματα για την περάτωση της συζήτησης αυτής. Έχει λήξει λοιπόν η συζήτηση και θα γίνει Πολύ σύντομα η ψηφοφορία. Διακόπτω για λίγα λεπτά την Σύνοδο Ολομέλειας.